Okay, I think we start, uh, and I'm happy to... Καλησπέρα. Χαίρομαι που βλέπω ότι έχουμε την Επίτροπο Μπιανκόφσκα εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά, εδώ και ένα χρόνο που συζητούσαμε το ίδιο θέμα, 14 Μαρτίου. Όχι, δεν είχαμε τις ειδούς του Μαρτίου, θα ήταν επικίνδυνο, 14 Μαρτίου. Την περασμένη φορά ήταν καρποφόρα η συζήτηση. Ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και αυτή τη φορά. Να σας πω ότι έψαχνα στο Google και διάβασα τις πολωνικές εφημερίδες τι λέγανε για την Επίτροπο Μπινκόφσκα και είδα κάτι που μ' άρεσε που γράφανε. Δεν είμαι Yorkshire Terrier, δεν είμαι ούτε Bull Terrier, δεν είμαι δεν είμαι ούτε πολύ καλή, αλλά ούτε η πολύ άγρια και καταπιστική. Επίτροπε Μπιενκόφσκα, είναι χαρά μας που είσαστε εδώ. Έχετε ένα δεκάλεπτο και μετά θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω θα με βρείτε καλή. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, σας είπε και ο Πρόεδρος, χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας σήμερα, ανταλλάξουμε απόψεις. Θέλω να σας ακούσω. Σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο σκάνδαλο Diesel πριν από ένα χρόνο σας ενημέρωσα για την πρόοδο που επετεύθη εφαρμόζοντας τις συστάσεις της Επιτροπής ΕΜΙΣ πέρσι τον Οκτώβριο. Σας υπέβαλα και την έκθεσή μας για τις σχετικές δράσεις που ακολούθησαν τις συστάσεις. Σας έδωσα και τις εκθέσεις των κρατών μελών που απεικονίζουν την κατάσταση των κρατών μελών. Είναι σημαντικότατο αυτό. Αλλά στο όλο δράμα είναι η βασική ηθοποίη τα κάτι μέλη. Συνεργαστήκαμε, να το θέσω έτσι. Εντατικά συνεργαστήκαμε από το Δεκέμβριο του 2015. Ελπίζω ότι παρατηρήσατε ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να αντιμετωπίσω τις συνέπειες του Dieselgate του σκανδάλου με τους κινητήρες diesel και κάτι εξίσου σημαντικό να αποφύγουμε κάτι τέτοιο να επαναληφθεί στο μέλλον. Συνεργαστήκαμε στενά μαζί σας με το Συμβούλιο προσβελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα οχήματα, τα μηχανοκίνητα. Κάναμε πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι θεμητό να το πει κανείς αυτό. Πολλά απομένουν να επιληθούν και θα πρέπει να ασκήσουμε και κάποια αυτοκριτική και εγώ ίδια αλλά ε, έχουμε ένα πιο αποδοτικό σύστημα εγκρίσεων με ανακλήσεις, δοκιμές των οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επίσης καταρτήσει και κανόνες για τις δοκιμές, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος βάσει της διαδικασίας ε, της νέας για την έρευνα και ανάπτυξη και το RTLP ένα παράδειγμα. Χάρη στο RDE, η πρόσφατη γενιά των διζελοκίνητων οχημάτων, μεταξύ 20 και 60 μιλιγκράμμ ε, οξυδίων του αζότου εκπέμπουν ανά χιλιόμετρο. Πριν ήταν περίπου 700 με 800 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Πιστεύω ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι πολύ καλό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Έχουμε το επίκαιρο θέμα της αποφάσεις του δικαστηρίου για το RDE. Θα σε εξηγήσω. Και στο Συμβούλιο αναφέρεται αυτό, αναφέρθηκε αυτό. Στην συνεδρίαση με την Επιτροπή, Έμι, θα ανακοινώσω το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα. Μέχρι τώρα έχουμε ανοίξει 8 διαδικασίες επί παραβάση. Έχουμε βελτιώσει τη διαφάνεια όσον αφορά τις ανακλήσεις οχημάτων στα κράτη-μέλη. Θέλουμε να αυξήσουμε και την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών εναρμονίζοντας την διαδικασία συλλογικής αποζημίωσης και προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε μια έρευνα για συνεργασία μεταξύ γερμανικών ε, αυτοκινητοβιομηχανιών, ούτως ώστε να καθυστερήσει κάπως η εγκατάσταση των διαφόρων συστημάτων για τη μείωση των εκπομπών. Έχουμε διάφορες προτάσεις, αλλά όπως σας είπα εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Δεν πρέπει να σταματήσουμε σε αυτό το στάδιο. Να σας πω και κάτι άλλο. Ε, είχαμε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και έλεγε ότι τα κράτη-μέλη δεν επέβαλαν καμία κύρωση στου κατασκευαστέ για παραβίωση του κανονισμού για έγκριση τύπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι τι κυρώσει δεν έχουν προβλεφθεί, δεν έχουν επιβληθεί. Ήταν, αλλά θα επιβληθούν σαν αποτέλεσμα της δικαστική διαδικασία, αλλά όχι από τι κυβερνήσει των κρατών μελών. Σχετικά με τι ανακλήσει των οχημάτων και οχήματα μη συμμορφούμενα, εκεί η κατάσταση δεν είναι ακόμα ικανοποιητική. Υπήρξε πρόοδος. Θα ξέρετε ότι πριν από ένα έτος ξεκίνησε η πλατφόρμα για τις ανακλήσεις. Ε, το μέσο ποσοστό ανακλήσεων αυξήθηκε από μέσο όρο 72 σε 79, αλλά 7 χώρες, τις κατονομάσω Βουλγαρία, Κροατία, Λετωνία, Μάλτα, Πολωνία, Ρωμανία, Σλοβακία εξακολουθούν να έχουν ποσοστά ανάκλησης κάτω από το 60%, πολύ χαμηλό ακόμα δεν ε, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δεν αυξάνεται το ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου 1,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα, διζελοκίνητα, που θα πρέπει κατεπηγόντως να ε, εξυγχρονιστούν. Και αυτό πέραν των παλαιότερων οχημάτων που ρηπαίνουν σημαντικά για τα παλαιότερα οχήματα, θα πρέπει να, γίνει, να υπάρξουν ανασκευές αυτών, ε, εγκατάσταση διαφόρων συστημάτων και μόνο μερικά κράτη-μέλη το κάνουν αυτό. Δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που έδωσε ένα εκατομμύριο ευρώ για πιλωτικά προγράμματα για τις δοκιμές εγκατάστασης των διαφόρων συστημάτων στα παλιά οχήματα. αλλά θέλουμε περισσότερη προσπάθεια, διότι παραδέχομαι ότι υπάρχει μεν μια αλλαγή όσον αφορά την προσέγγιση και στα κράτη-μέλη και στη βιομηχανία, αλλά Χρειαζόμαστε περισσότερη προσπάθεια από τα κράτη-μέλη και περισσότερη προσπάθεια από τη βιομηχανία μας. Διαφορετικά όλες οι προσπάθειές μας θα είναι εις Η βιομηχανία θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και όπως επαναλαμβάνω πρωτίστως είναι προς δικό τους όφελος το μέλλον. Αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να είναι πολύ πιο δραστήριες. Βλέπω πρόοδο, είναι ασύγκριτη κατάσταση εν συγκρίση με τη δική μου εμπειρία του 2015 και του 2006 και σε σύγκριση με τώρα, αλλά πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν. Έχουμε καινούριε συσκευέ που ανακαλύπτονται, που παρακάμπτουν τα συστήματα μειώσεων των εκπομπών και πρέπει να πω ότι η βιομηχανία είναι αργή όσον αφορά την εφαρμογή της ηλεκτρικής κινητικότητας ή βιώσιμη βιώσιμης κινητικότητας. Με τα νέα πρότυπά μας για το δίξιο του άνθρακο τους ταρακουνήσαμε, αλλά μόνο λίγες αυτοκινητοβιομηχανίες ανοιχτά έχουν ε, συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τα διπλώματα ευαισθητεχνίας σε αυτό το τομέα. Αλλά είναι βασική τεχνολογία που θα μειώσει την εκπομπή άνθρακο και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη. Θέλουμε πραγματικά να αναπτύξουμε ε, μία λυσίδα αξία για τις ε, μπαταρίες στην Ευρώπη ε, και ελπίζουμε να μην χάσουμε την ευκαιρία. Σχεδιάζουμε να δώσουμε πολλά χρήματα σε αυτόν τον τομέα, διότι είναι εκ των ουκ άνευ για μας, αν θέλουμε αυτό το τμήμα της κινητικότητας να αναπτυχθεί. Τώρα, όπως σας προανέφερα, πρέπει να κοιτάξουμε με κριτικό όμα τα πεπραγμένα και για τη γενική απόφαση του δικαστηρίου. Πριν από δύο μήνες βγήκε στις 13 Δεκεμβρίου και αποφάσισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπέρασε τα όρια των εξουσιών όταν υιοθέτησε τους παράγοντες συμμόρφωσης με τον κανονισμό RD και βέβαια πρέπει να αντιδράσουμε όσον αφορά αυτή την απόφαση. Θέλουμε να δώσουμε στο Κοινοβούλιο πιο ενεργό ρόλο, ισχυρότερο ρόλο. Δεν θέλω να δικαιολογήσω ή να... Θα ήθελα να, εξηγήσω κάπως την όλη κατάσταση. Ευτυχώς όλοι μας αυτή την αίθουσα πριν από 3,5 χρόνια είμαστε στο Κοινοβούλιο και το συζητήσαμε και εγώ παρουσίασα το θέμα. Θυμόμαστε τις, τη ζωηρή συζήτηση και την κατεπίγουσα ανάγκη που υπήρχε να βρεθεί μια λύση. Και γι' αυτό πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Και επανειλημμένως είπα ότι πρέπει και εγώ να κινηθώ, να δραστηριοποιηθώ, να αναλάβω τις ευθύνες μου. Σήμερα δυστυχώς, παρόλο που δεν αφισβήτησε το δικαστήριο τους παράγοντες συμμόρφωσης αυτούς καθ' αυτούς, αλλά τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, σήμερα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε νέα πρόταση νομοθετικού περιεχομένου στα πλαίσια της συναπόφασης. Θα θυμόσαστε ότι το δικαστήριο μας έδωσε μόλις ένα χρόνο, μόλις. Κανονικά χωρίς εκλογές, εντάξει θα ήταν, θα αρκούσε το χρονικό διάστημα. Θα μπορούσαμε να διεκπαιρεώσουμε το έργο μας αλλά υπό τις παρούσες ε, περιστάσεις νομίζω ότι είναι στενά τα χρονικά περιθώρια. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ε, υποβάλει έφεση όσον αφορά την απόφαση. Οι εμπειρογνώμονές μας, οι νομικοί, λένε ότι υπάρχει βάση για τέτοια έφεση. Δεν θέλω όμως να με παρεξηγήσετε, να παρερμηνεύσετε. Εγώ εστιάζομαι στο να θεσπίσουμε εγκαίρως την κατάλληλη νομοθεσία και θέλω εσείς το Κοινοβούλιο να έχετε λόγο σε αυτό. Πρέπει για μία ακόμη φορά να είμαστε δίκαιοι, να είμαι δίκαιοι. Έχουμε μόλις ένα χρόνο, χρόνο εκλογών και θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει πρόβλημα. Θα επηρεάσουμε την παραγωγή εκατομμυρίων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 24 Φεβρουαρίου του 2020 θα ακούσουμε τι έχει να πει η βιομηχανία. Η βιομηχανία θα μας πει ότι είναι το τέλος του κόσμου που έφτασε για αυτούς, ότι θα μας απειλήσουν ε, οι απώλειες θέσεων εργασίας. Και εγώ και εσείς το έχουμε συνηθίσει αυτό να το ακούμε. Πραγματικά εγώ ανησυχώ για την αντίδραση των πολιτών, την αντίδραση της κοινωνίας. Εσείς τους ακούτε καλύτερα από μένα, έχετε περισσότερη επαφή με αυτούς από ότι εγώ, παρόλο που και εγώ έχω επαφή με τον κόσμο. Ίσως πει ο κόσμος ότι για όλα αυτά φταίνε οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες των Βρυξελών που δεν έχουν εφαρμόσει τα σωστά μέτρα. Αυτό που είναι σημαντικό πιστεύω για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι να αποφύγουμε μια επανάληψη του φαινομένου και να εστιαστούμε στο μέλλον. Προπαρασκευαστική εργασία για μελλοντικά πρότυπα για τι εκπομπέ είναι κάτι που ήδη έχει δρομολογηθεί στην Κραϊόβα τον επόμενο μήνα. Η Ρουμανική Προεδρία διοργανώνει μία διάσκεψη έναν οδικό χάρτη προς καθαρά οχήματα. Αυτό είναι ένα από τα θέματα συζητήσεως. Σαν αντίδραση στην απόφαση του δικαστηρίου ετοιμάζουμε νέα νομοθεσία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και θα είμαι εδώ μέχρι την τελευταία στιγμή της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τον Οκτώβριο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρξει αυτή η νομοθεσία. Ταυτόχρονα, πιθανότατα θα υποβάλουμε έφεση Εν είδη συμπερασμάτων από κάποια πράγματα. Όπως πάντα μπορείτε να βασίζεστε σε μένα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά βέβαια για να κάνουμε ουσιαστική διαφορά πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και η βιομηχανία όπως σας είπα θα συνεχίσω την προσπάθειά μου μέχρι την τελευταία ημέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου εμφάνιση μπροστά σας σαν Ευρωπαία Επίτροπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που κάναμε μαζί. Χωρίς την υποστήριξή σας δεν θα τα πετυχαίναμε αυτά. Ψηφίσατε επίσης τους παραγόντες συμμόρφωσης, παρόλο που εκφράσατε τότε ανησυχίες για τη διαδικασία, αλλά από τη δική μου πλευρά μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να κινηθούμε τόσο γρήγορα όπως κινηθήκαμε. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω να ακούσω τις αντιδράσεις σας και να συζητήσουμε, να ακούσω ερωτήσεις και να απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στον πρώτο κύκλο ερωτήσεων. Έχετε δύο λεπτά και θα ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ. Και την κυρία Κώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την παρουσίασή σας και εν γέννη για την προσπάθεια που καταβάλλατε σε αυτό το χαρτοφυλάκι όπως και στα άλλα θέματα με τα οποία ασχολείστε. Από την αρχή του Dieselgate δείξατε ότι θέλετε να προσπαθήσετε να βρείτε λύση και να συνοδεύσετε και, και το έργο της Ερευνητικής Επιτροπής και να ετοιμαστεί κατάλληλη η έκθεση που παρουσιάσει τα διάφορα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Είπατε ότι επετεύχθη πρόοδο, ούτω ώστε αυτή η απαράδεκτη απάτη που γνωρίσαμε για του κινητήρε δίζελ να μην επαναληφθεί. Αλλά μα είπατε επίση ότι ακόμα υπήρχαν πολλά που πρέπει να γίνουν. Μα εξηγήσατε ότι έλεγχο των εκπομπών ενισχύθηκε με νέε διαδικασίε ε, των δοκιμών. Και όλα αυτά οδηγούν σε μια ευρωπαϊκή ρύθμιση ε, πιο αυστηρή. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτά τα μέτρα υιοθετήθηκαν με τεράστια ταχύτητα, διότι αυτό ήταν αναγκαίο, ήταν απαραίτητο, αλλά ταχύτητα η οποία περιέπλεξε το, το έργο των κατασκευαστών. Εκεί έχουν πιο μακροσκελείς και χρονοβόρους κύκλους παραγωγής και δεν έχουν το χρόνο να προσαρμόσουν κατάλληλα τα οχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να λησμονήσουμε τις ψευδείς καλές ιδέες που μας κάνουν να θυσιάσουμε τον δίζελ υπέρ της βενζίνης, που ή να πάμε προς τα χήματα με μηδενικές εκπομπές που απολογισμός τους ε, όσον αφορά τον άνθρακα δεν είναι τόσο αθώος όσο φαίνεται από πρώτη ματιά. Ερωτήσεις. Το Σεπτέμβριο του 2018 ένα πρώτο βήμα του τεστ RDE εφαρμόστηκε. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τις συνέπειες, τα αποτελέσματα, όσον αφορά το στόλο των κατασκευαστών. Συγκράτησε αυτό που είπατε, ότι ακόμα υπήρχαν κάποια, κάποια μηχανισμοί ε, που υπερκεράζουν, μπορούν να υπερκεράσουν. Τι γίνεται με τεχνολογία την υβριδική. Μπορείτε να μας πείτε πού βρίσκεται η τεχνολογία πλευράς των κατασκευαστών και ποιος είναι ο βαθμός προσαρμογής ε, στις νέες διαδικασίες δοκιμασιών. Ε, μπορείτε πραγματικά να προσμετρήσετε τις συνέπειες, τα αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Καθήν Βαν Πρέμπτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε. Ε, με στεναχωρεί που άκουσα ότι είναι η τελευταία φορά που έρχεστε. Μπορείτε να επιστρέψετε. Αλλά ας ξεκινήσω ε, αναφερόμενοι όχι σε αυτά που έγιναν στο παρελθόν, αλλά λέγοντας ότι είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που κάναμε στην Επιτροπή εμείς και το καλό αποτέλεσμα, δηλαδή τη φιλόδοξη έκθεση την οποία υπερψηφίσαμε. Να πω επίσης ότι η ανάλυση της Επιτρόπου μας βρίσκει σύμφωνους. Έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό και σε επίπεδο κρατών ε, μελών αλλά η αξιολόγηση είναι αρνητική για να μην πω τραγική. Επίσης, δεν υπάρχει και δυνατότητα αλλαγή προ το παρόν. Υπάρχει έλλειψη βούληση. Αλλά να πω καταρχά πω, ε, κύριε Επίτροπε, με απογοητεύει το γεγονός ότι ότι θα προχωρήσετε σε έφεση για την απόφαση του δικαστηρίου ε, σχετικά με τον ε, παράγοντα συμμόρφωσης. Εκείνη την εποχή ήδη είχαμε πει πως κάτι τέτοιο δεν είναι δημοκρατικό. Έχει έχουν λοιπόν αλλάξει οι κανόνες ε, στην πορεία και χρησιμοποιείται μία μεθοδολογία η οποία ε, δεν είναι αποδεκτή, δεν πρέπει να είναι αποδεκτή. Αυτή ήταν η απόφαση του δικαστηρίου και εγώ θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να κρατήσετε, ε, να παραμείνετε στην καλή θέση στην οποία είστε, να συνεχίσετε την καλή δουλειά με το Euro 7 να υποβάλλεται μία πρόταση τόσο για το γύρο 7 όσο και για, την, ε, για τις απαιτήσει συμμόρφωσης. Έπειτα. Και μία άλλη ερώτηση σχετική με αυτό. Στην Επιτροπή εμείς υπήρχαν πάντα ανησυχίες ε, για το αν οι καταναλωτές αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στους καταναλωτές της, ε, των ΗΠΑ και στους καταναλωτές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές και ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα οχήματα που αγοράστηκαν στη Γερμανία είπατε ότι για να γίνει μετασκευή όχι μόνο στο λογισμικό αλλά και στο υλικό μέρος ε, πρέπει να ε, επιδοτηθούν τα οχήματα και πρέπει να καθαρίσει ο στόλος. Όμως, κυρία Επίτροπε, γιατί στα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν θα δοθούν ε, επιδοτήσεις, δεν θα έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να καθαρίσουν τα αυτοκίνητά τους να, και πλέον καθαρό ντίζελ έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη πλέον στα καθαρά οχήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φροντίσετε να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεμεσμέκερ έχει το λόγο από την ομάδα ICR. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει ως τώρα. Η Κάθλιν Βαν ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής εμείς, εγώ ήμουν ένας από τους αντιπροέδρους, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι σίγουρα το Dieselgate δεν έχει τελειώσει, δεν το έχουμε αφήσει πίσω μας. Και έχω μερικές ερωτήσεις από την πλευρά μου. Πρώτον, η απόφαση του δικαστηρίου. Όπως είπε και η Καθλίν, υπάρχει δυνατότητα άσκησης έφεσης και αυτή είναι και η πρόθεσή σας. Όμως θεωρώ πως θα στείλουμε ένα λάθος μήνυμα με την πράξη αυτή, ιδιαίτερα εν ώψη ευρωεκλογών. Ίσως κάποιοι από εμά δεν επιστρέψουν, θα διακοπούν είναι οι εργασίες μας σίγουρα και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την ταχύτητα που έχουμε μετά τις εκλογές. Έπειτα, το ελεκτικό συνέδριο στο οποίο αναφερθήκατε δημοσίευσε ένα ενημερωτικό έγγραφο. Αλλά δεν μου φαίνεται πως τα στοιχεία που περιέχει είναι πλήρη. Η κυριότερη πρόκληση είναι ο έλεγχος ε, καταλληλότητας ε, της αγοράς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη στο να το εφαρμόσουν. Θα υπάρχει δυνατότητα για τους ε, κατασκευαστές να μειώσουν τις εκπομπές και ταυτόχρονα να διεξάγουν τους ε, ελέγχους ε, καταλήλωτο αλλά και τους ελέγχους εκπομπών ε, οξυδίου του αζότου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνει από ένα τρίτο μέρος και θα πρέπει ταυτόχρονα να φροντίσουμε να μειωθεί το οικονομικό κόστος αυτών των ελέγχων. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα. Πάντα σε συνεργασία με τα κρατημέλη βέβαια. Επίσης είπατε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία με τα κρατημέλη. Τι λοιπόν προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό. Πώς θα μπορέσετε να δώσετε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Διότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τα κράτη-μέλη και εκείνα να συμμορφωθούν με τις ε, αντίστοιχες ε, οδηγίες ε, για τον έλεγχο Η δική σας Γενική Διεύθυνση και η Γενική Διεύθυνση για περιβαλλοντικά θέματα, τι προτίθεται να κάνουν. Ρωτάω ως πρώην δημοσιογράφος και έχω και ειδικό ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου των φιλελευθέρων, ο κύριο Κερμπράντι έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Η πρώτη ερώτησή μου είναι πιο πολύ ερώτηση επί της διαδικασίας και της διοργανικής συνεργασίας. Η απάντηση στην πρώτη επίσημη ερώτηση είχε τη μορφή προσωπικής επιστολής ε, στον πρόεδρο της Επιτροπής ΕΜΙΣ και όχι επιστολή από τον, πρόεδρο της Κομισιόν, από τον ε, Γενικό Γραμματέα της Κομισιόν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν επίσης, ε, όχι μόνο αυτό, αλλά και το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιόρισε την απάντησή της σε συγκεκριμένα θέματα και δεν απάντησε σε όλα. Ε, δεν απάντησε σε ερωτήσεις για κακοδιοίκηση, για παράκαμψη κανόνων, ε, στα συμπεράσματα. Καμία αντίδραση λοιπόν σε αυτό το θέμα. Επίσης μου έκανε έκπληξη το εξής. Στην απάντησή σας ε, είπατε για ορισμένα θέματα ότι δεν μπορείτε να πατήσετε διότι ε, δικαίωμα απάντηση ε, και αρμόδιο για να απαντήσει είναι μόνο ο Γενικό Γραμματέα, ο πρόεδρο τη Κομισιόν. Πώ λοιπόν γίνεται να μην απαντάτε σε ορισμένα σημεία γιατί δεν είστε αρμόδια, γιατί αρμόδιο είναι ο πρόεδρο Κομισιόν. Ε, είχα την εντύπωση ότι η απάντησή σα είναι η επίσημη απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή λοιπόν η αναπάντηση προς την Επιτροπή έμιση είναι προσωπική σας απάντηση, μιλάτε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τι είναι. Επίσης, ε, σε ό,τι φορά την ε, έφεση που θα σκηθεί, αυτό είναι δική σας απάντηση ή μιλάτε πάλι εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, είναι γεγονός ότι τόσο εσείς όσο και εμείς έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά για να παρουσιάσουμε καινούργια νομοθεσία, όμως το πιο δύσκολο έργο είναι να καθαρίσουμε αυτό το χάος και αυτή τη, αυτά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Να καθαρίσει λοιπόν το τοπίο. Βλέπουμε ότι η Γερμανία θα διοργανώσει την ε, διάσκεψη για τον ντίζελ, ίσως αποζημιώσει ε, καταναλωτές οι οποίοι είναι κάτοχοι τέτοιου αυτοκινήτου, αλλά τα αυτοκίνητα τι θα απογίνουν, θα πουληθούν σε μια άλλη χώρα και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στους δρόμους. Πού είναι λοιπόν η ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα αυτό. Κατανοώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νομικούς περιορισμούς, όμως πολιτικά είναι πολύ πιο εύκολο να αναλάβετε ηγετικό ρόλο. Και αυτό που θα περίμενα από τον πρόεδρο της ε, Κομισιόν, ιδιαίτερα ως αντίδραση στο μεγαλύτερο βιομηχανικό σκάνδαλο των τελευταίων ετών, είναι ε, να αναλάβει την πρωτοβουλία. Γι' αυτό λοιπόν εσείς τι έχετε να πείτε για την έλλειψη αυτή πρωτοβουλίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπάς Άικουτ έχει το λόγο εξ ονόματος των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Να πούμε καταρχάς ότι οι απαντήσεις σας ε, στα συμπεράσματα και τις συστάσεις ήταν σχεδόν οριακές, σχεδόν ανεπαρκείς. Ε, λείπει η ουσία. Ε, ενώ αντίθετα ακούστηκαν σοβαρές ε, κατηγορίες κατά της Κομισιόν. Θέλουμε όχι μόνο να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον, αλλά να μάθουμε τι πραγματικά συνέβη. Το γεγονός είναι επίσης ότι συνεχίζουν να κυκλοφορούν βρώμικα ε, οχήματα που καίνε ντίζελ στο δρόμο. Μας είπατε για κάποια εκατομμύρια, 16 ε, εκατομμύρια όμως έχω ακούσει από άλλες πηγές ότι είναι πάνω από 40 εκατομμύρια. Εσείς τι στοιχεία έχετε να μας δώσετε. Πρόκειται μόνο για οχήματα της, ε, του ομίλου Volkswagen, διότι ακούγεται ότι υπάρχουν και άλλες ε, εταιρείες που έχουν εξαπατήσει τους ε, καταναλωτές. Πού είναι η ηγετική ικανότητα και ο ηγετικό ρόλος της Κομισιόν. Εσείς μπορείτε να προτείνετε συγκεκριμένες κατευθυντήριε γραμμές στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να βελτιώσουν το σύστημα ε, ανάκλησης και μετασκευής των ε, οχημάτων. Σίγουρα είναι εθνική αρμοδιότητα αυτό το θέμα, όμως εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορείτε να ανεβείτε και να αναλάβετε ηγετικό ρόλο, να, καθοδηγήσετε. Δεν αρκεί να λέμε στους πολίτες ε, λόγια, διότι οι πολίτες έτσι καταλαβαίνουν ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικαστήριο, μου θυμίζει μια περίπτωση στις κάτω χώρες όπου το δικαστήριο απεφάνθη και ε, η Ολλανδική πλευρά απάντησε ότι εντάξει θα σεβαστούμε την απόφαση αλλά ναι και όχι κιόλα, γιατί μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Τι έγινε τελικά στην ε, πράξη. Ε, άσκησαν έφεση στην απόφαση, έχασαν πάλι, αλλά στην πράξη δεν έγινε τίποτα. Και βλέπω πως και εσείς προς αυτήν την κατεύθυνση πάτε, θα κινηθείτε νομικά χωρίς να γίνει τίποτα ουσιαστικό. Μας είπατε επίσης ότι θα υποβάλλετε πρόταση, ότι αυτή είναι η επιθυμία σας. Ε, τι πρόταση είναι αυτή, θέλω να ρωτήσω εγώ. Διότι, να σας το πω ευθέως, δεν χρειάζομαι πρόταση. Το δικαστήριο απεφάνθη. Αν θέλουμε να χαμηλώσουν τα στάνταρ σε σχέση με το 2009, πρέπει να ακολουθήσουμε ε, την ε, συνήθεια διαδικασία. Εμείς ε, είχαμε ενστάσεις, χάσαμε, αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουν τα στάνταρ. Εμείς θέλουμε να παραμείνουν όσα έχουν. Δηλαδή, τι, τι μας λέτε, ότι θα υποβάλλετε πρόταση για να αλλάξουν τα πρότυπα για να χαμηλώσει το επίπεδο. Αυτό είναι το μήνυμά σας προς τους Ευρωπαίους πολίτες, ότι ναι, θα χαμηλώσουμε τα πρότυπα και θα πάμε προς πιο βρώμικο αέρα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Εξανόματο της Γκουε ή κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι χτες αργά το βράδυ, ίσως και νωρίς το πρωί, Είπατε πως εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνήσαμε έναν κανονισμό ο οποίος θα θέσει τους κανόνες για τα νέα βαρέα οχήματα και ότι αυτό έκλεισε το νέο πλαίσιο για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε όλα τα οχήματα και αυτά θα συμπεριλάβουν και τα οχήματα με εναλλακτικούς κινητήρες. Αυτό λοιπόν ε, υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να παρακολουθούμε τις εκπομπές έτσι ώστε να μην ξανά έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Γνωρίζουμε όμως όλοι πολύ καλά πως ε, ενώ το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, αυτό που πετύχαμε δεν είναι αρκετό από μόνο του. Η αυτοκινητοβιομηχανία μετακινείται προς εναλλακτικά καύσιμα και οι ηλεκτρικούς κινητήρες. Το πακέτο της καθαρής κινητικότητας, για παράδειγμα, εκεί τονίσαμε πως θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλο τον κύκλο ζωής των οχημάτων, έτσι ώστε να πετύχουμε την ισορροπία στην αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσει πως δεν θα επαναλάβουμε το παρελθόν με την πρώτη γενιά των βιοκαυσίμων. Θα πρέπει λοιπόν να περιγράψουμε τι είδους εκπομπές και σε ποιο ύψος θα μπορούν να εκπέμπονται από τα, εναλλακτικά, τα με εναλλακτικά κινητήρα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα ηλεκτροκίνητα από τη στιγμή της κατασκευής μέχρι και της ανακύκλωσης. Το είπατε κι εσείς, η παραγωγή, ε, για παράδειγμα, και η καταστροφή των, ε, της μπαταρίας ε, στα ηλεκτροκίνητα είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε εξετάσει καθόλου και υπάρχουν κάποια αρνητικά εξωτερικά στοιχεία για τα ηλεκτροκίνητα, τα οποία αυτή τη στιγμή αμελούμε μεταφέροντας το πρόβλημα στις τρεις χώρες. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να κυλήσει έτσι, γιατί θα επαναλάβουμε τα προβλήματα που είχαμε για παράδειγμα με το φινικέλαιο. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα υπονομαζόμενα καθαρά οχήματα και να έχουμε τον ε, κόσμο ε, τον υπόλοιπο να υποφέρει ε, σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση που αυτή μας την επιλογή. Τι θα κάνετε λοιπόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναλύσετε όλα αυτά τα νέα οχήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Και επίσης πείτε μου, τι θα κάνετε πιο συγκεκριμένα προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα αφενός ε, που αντιμετωπίζουμε και άλλα προβλήματα φετερού τα οποία αναδύονται και ακόμα δεν έχουμε περιγράψει. Ωραία, λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στην Ελεονόρα Εύη από το CFTD. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Επίτροπε. Σημαντική αυτή η συζήτηση σήμερα, διότι στο Ευρωκοινοβούλιο πιστεύω ότι οι φωνές των συναδέλφων δείχνουν ότι ερμηνεύουμε ε, κάπως ε, με ανήσυχο τρόπο το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια, ε, κάπως βρίσκουμε λύσεις με τα έγγραφα που μπροστά μας, την απόφαση του ΔΕΚ, και την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Και τα δύο αυτά έγγραφα που έχουν εμβαθύνει, μας λένε το Ευρωκοινοβούλιο, πάντα είχε δίκιο, που προσπιζόταν μια θέση σαφή, όπως τους παράγοντες συμμόρφωσης. Και εγώ ανήκω σε αυτούς που πολέμησε για να αποφύγουμε να θεσπιστούν αυτοί οι κανόνες, αυτοί οι παράγοντες συμμόρφωσης. Δεν πέτυχαν τίποτα επέτρεψαν προς τους κατασκευαστές να εξακολουθούν ε, να ε, ξεπερνάνε τα όρια ε, που είχαν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σοβαρό, πολύ σοβαρό που σήμερα είμαστε στην ίδια κατάσταση. Σας ερωτώ κύριε Επίτροπε, υπό το φως της εκθέσεως και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που μας λέει ότι υπάρχουν ανεπαρκείς διατάξεις όσον αφορά την ταξινόμηση στην Ευρώπη. Ανεπαρκές το πλαίσιο και οι προδιαγραφές για να έχουμε πραγματική μείωση των εκπομπών. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση και η έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τα χήματα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν και που θα έπρεπε να αποσυρθούν ε, είναι κάτι που μας δίνει απλώς ένα κομμάτι της όλης εικόνας που, που δείχνει το συνολικό πρόβλημα. Και κάτι άλλο αυτό. Της ε, αναδρομικής μετασκευής των οχημάτων. Σε κάποια κάτι μέλη εθελοντικά γίνεται απόσυρση παλαιών οχημάτων, όπως στην Ιταλία. Κάναμε αποσύρσεις εθελοντικές. Αλλά υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά και hardware και software. Υπάρχουν διαφορές. Έχετε προβλέψει πρωτοβουλίες για να μπορούν να εξυγχρονιστούν τα οχήματα που σήμερα κυκλοφορούν και να μπορέσουν να γίνουν να μειώσουν τις ρηπαντικές ε, ουσίες που εκπέμπουν και να μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς να παραβαίνουν τις διατάξεις. Δεν έχουμε κάποιο με το ΙΕΝΕΦ. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει. Δεν υπάρχουν λοιπόν τερίε Yorkshire που να είναι συμπαθητικά. Τα πιο συχνά που συναντάμε είναι τα Bull Terrier, οπότε αυτό το αφήνω εκεί και σας προτείνω να απαντήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Να σας πω πως ε, πάντα ο τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα. Όμως και από τις δικές σας ε, παρεμβάσεις κατάλαβα πως τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε κάνει καλή δουλειά. Δυστυχώς, όπως πήγε αρκετές φορές, αλλά ίσως και εδώ υπάρχει κάποια θετική πτυχή, το σκάνδαλο με τον Ντίζελ μας βοήθησε και προχωρήσαμε γιατί με την προσέγγιση που είχα δει και την είχατε δει κι εσείς, κυρίως με την βιομηχανία, δεν θα είχαμε προχωρήσει τόσο γρήγορα και το λέω δυστυχώς γιατί από τις συναντήσεις που είχαμε τους εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν πάρα πολύ σκληροί και τα πρώτα δύο χρόνια δεν ήταν καθόλου συμπαθητικοί και μετά άλλαξαν γιατί είδαν πως η κοινωνία η ίδια αλλάζει και απαιτεί από αυτούς να αλλάξουν προσέγγιση, να αλλάξουν πολιτική για να προχωρήσουν σε πιο, καθαρά, πιο καθαρή παραγωγή και πιο καθαρά οχήματα. Δεν πιστεύω πως η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν γνώριζε τόσα χρόνια ότι πρέπει να αλλάξει. Αλλά Εντάξει, είχαν βολευτεί, δεν έκαναν τίποτα, γιατί δεν είχε συμβεί τίποτα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει σχέδια. Ή το μερίδιο που έχει κανείς ε, στις εκπομπές από τη μία μέρα στην άλλη, από το ένα εργοστάσιο ε, στο άλλο. Έτσι, μειώντας 30-40% αυτή ήταν η κατάσταση τώρα για την έφεση για την ένσταση και αυτή είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσω ίσως έτσι στον κύριο Γκαμπράντη εγώ εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όποια επιστολή υπογράφω εκπροσωπεί αποτελεί την επίσημη απόκριση της Ευρωπαϊκής Επιστολής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πρόεδρο της Επιτροπής ΕΜΙΣ. Η απόφαση των Επιτρόπων ήταν να υποβάλουμε ένσταση και το λέω προσωπικά, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να έχουμε την νομοθεσία έτοιμη μέσα σε τούτη τη χρονιά. Και αν η έγκριση της νέας νομοθεσίας γίνει μέσα στα χρονικά θόρια μπορώ να αποσύρω αυτή τη ε, διαδικασία έφεσης οποιαδήποτε στιγμή και αυτό αποτελεί δική μου προσωπική δέσμευση αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα φέτος όταν ο χρόνος ε, μας πιέζει και έχουμε μέχρι τις 20 τόσο Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς γιατί μπορεί να βρεθούμε να μην έχουμε τίποτα νομοθετικά ομιλώντας στη διάθεσή μας. Δεσμεύομαι λοιπόν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η πρώτη μας προτεραιότητα και η πρώτη λύση είναι νέα νομοθεσία. Εάν όμως, επειδή είναι δύσκολη χρονιά και το ξέρετε, γιατί από τα μέσα Μαΐου μέχρι και μερικούς μήνες μετά δεν θα είμαστε εκεί για να κλείσουμε με το θέμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πώς θα είναι το καινούργιο κοινοβούλιο. Αυτή λοιπόν είναι η ασφαλιστική μας δικλίδα για το συγκεκριμένο σημείο. Για τα αποτελέσματα της, ε, των πρώτων δοκιμών, να σας πω ότι ήταν πολύ θετικά και όλα τα οχήματα τα οποία έχουν περάσει αυτή την ανεξάρτητη δοκιμή είναι, συμμορφούνται. Και επειδή η ερώτηση έχει να κάνει με το τι είδους νομοθετική πρόταση θα υποβάλουμε, εμείς θα έχουμε τους ίδιο, τα ίδια σημεία, α, σημεία συμμόρφωσης 2,1, 1,43, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Εμείς κάναμε και την ετήσια ε, αναθεώρηση του τεχνικού περιθωριού πέρσι και καταλήξαμε σε κάτι χαμηλότερο από το 1,43 που είναι στη θέση του 1,5 και συνεχίζουμε ακόμα φέτος μαζί με τη σχετική επιτροπή για να κλείσουμε το θέμα ε, το δεύτερο εξάμεινο και έχουμε δεσμευθεί ε, με τη δήλωση που έκανα εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το τεχνικό περιθώριο να το περιόρισουμε μέχρι σχεδόν το 1 μέχρι το 2023. Ακολουθούμε λοιπόν αυτή την άριστη κατά τη γνώμη μου κατεύθυνση και πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Τα έχουμε και το νέο καθεστώς έγκρισης τύπου Είμαστε σε επαφές με τα κράτη-μέλη. Θα κάνουμε την πρώτη συνάντηση το Μάρτιο για να προετοιμάσουμε την ε, κοινή ε, απόκριση, γιατί θα είναι ε, μέσω της ε, Τεχνικής Επιτροπής που θα γίνει η προσπάθεια και νομίζω ότι και μέχρι τα τέλη της δικής μας θητείας θα έχουμε εγκρίσεις τύπου. Τώρα, για τους κατοίκους Γερμανίας που θα έχουν τα επιπλέον χρήματα για τα καθαρά οχήματα, γιατί δεν είναι Γερμανοί, είναι όσοι είναι κάτοικοι στη Γερμανία, να σας πω πως από την αρχή, πως τα κράτη-μέλη που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και που θεωρούν ότι είναι υπεύθυνα, αυξάνεται συνέχεια. Αλλά δεν είναι ακόμα ικανοποιητικό ο αριθμό. Με κάποια κράτη-μέλη δεν είναι εντάξει η σχέση μας στο σημείο αυτό, αλλά δεν είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα κατευθύνω αυτή τη συζήτηση και σε λίγο θα απαντήσω και για το θέμα της πολιτικής ε, ηγεσία από πλευράς Κομισιόν, αλλά υπάρχει τεράστια ευθύνη από τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη λογοδοτούν στους πολίτες τους. Τα πιο βρώμικα αυτοκίνητα στην Ευρώπη είναι στις χώρες που και η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι χειρότερη. Είναι ευθύνη των κρατών μελών. Αυτό. Και δεν έχουν αποκριθεί αρκετά. Δεν έχουν ανταποκριθεί αρκετά αυτά τα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμής. Για το θέμα της πολιτικής ηγεσία και του κατά πόσο δείχνουμε τέτοιου είδους ηγετικές ε, τάσεις θα γίνει μία διάσκεψη στο κράιο σε ένα μήνα περίπου. Και εκεί πιστεύω θα είναι κατάλληλη στιγμή για να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Γίνεται τακτικός διάλογος με τα κράτη-μέλη και έχουμε και γύρω τραπέζες για θέματα diesel σε πολύ τεχνικό επίπεδο και βασιζόμενοι στις απαντήσεις των κρατών μελών εμείς βλέπουμε ποιος θα είναι ο δικός χάρης που θα μας οδηγήσει στα καθαρά οχήματα που ε, συμπεριλαμβάνει κάποιο είδους ε, ε, οικοδομικά κατασκευαστικά μπλοκ που θα τα χρησιμοποιήσουμε για να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτά όλα τα απαραίτητα μέτρα to and και όλα αυτά για να εξασφαλίσουμε πως θα είναι καθαρό από ντίζελ το μέλλον. Στόχος μας είναι το σχέδιο αυτό και ο δικός χάρτης. Αυτός ο δικός χάρτης να εγκριθεί σε ένα μήνα στο Κράγιοβα. Και πιστεύω ότι καλό είναι να γίνεται αυτή η, η συνδιάσκεψη. Πάντα χρειαζόμαστε μια φορά το χρόνο να βλεπόμαστε σε επίπεδο ηγετών ε, κρατών ε, μελών και πρέπει να σου πω ότι την τελευταία φορά δεν ανταποκρίθηκαν όλοι όσο θα έπρεπε. Επίζω πως θα είναι εκεί για να εγκρίνουν και να εκινήσουν αυτόν τον οδικό χάρτη. Uh, on the, uh, on the guidelines. Για τις κατευθυντήριες γραμμές. Να πω δύο λέξεις το συζητήσαμε. Έχουμε κατευθυντικές γραμμές για διάφορα ε, μηχανήματα και πιστεύω στον οδικό χάρτη ένα από αυτά τα μέτρα που θα μας βοηθήσουν είναι αυτό το ποσό που θα πάει για το 1,6 εκατομμύρια Volkswagen που θα πρέπει να ανακληθούν για να αλλάξουν οι συσκευές. Και το είπα στην πρώτη μου παρουσίαση πως όλα αυτά θα γίνουν επιπλέον των εκατομμυρίων αυτοκινήτων μικροφόρου στους δρόμους που είναι ευρώμικα οχήματα. Και εδώ βέβαια θα πρέπει να αναλάβει το θέμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απαράλληλα είναι και πολύ σημαντικό θέμα για τα κράτη-μέλη και πρόβλημα για τις κυβέρνησεις τους και τις τους και γι' αυτό το επανέρχομαι. Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη αυτή με την απαραίτητη σοβαρότητα. Και υπάρχουν σημεία της Ευρώπης όπου ο αριθμός των βρώμικων αυτών οχημάτων είναι σε μεγαλύτερη πυκνότητα από ό,τι αλλού μετά των όσων πετύχαμε συλλογικά, γιατί αυτό πρέπει να το πω, έγκριση τύπου, νέο RDE, WLTP, όλα αυτά, ε, οι εκπομπές διοξιδίου για τα φορτηγά, όλα αυτά, αν τα συνδυάσουμε μεταξύ τους, βλέπουμε πως αν συμπληρωθούμε την καλύτερη προσέγγιση των ε, αυτοκινητοβιομηχανιών και με την καλύτερη προσέγγιση που ακολουθούμε εμείς, για να μην λέμε συνέχεια ότι θα χαθούν θέσει εργασία στο κλάδο, ε, να σα πω πω αν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει, θα καταστραφεί ο κλάδο ολόκληρο, όχι μόνο κάποιε θέσει εργασία. Γιατί χρειαζόμαστε να έχουμε καθαρή παραγωγή, καθαρά οχήματα και καθαρό αέρα στην Ευρώπη. Αν λοιπόν δεν τα κάνουμε όλα αυτά μαζί, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αλλά πιστεύω ότι έχουμε ήδη κάνει πρόοδο και πρέπει να το παραδεχτούμε και εσείς το παραδέχεστε, είναι κομμάτι της εντολής σας και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των όσων κάνετε εδώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Ξεκινάμε το ΕΛΚ. Δεν βλέπω να ζητούν μέλη του ΕΛΚ το λόγο. Υπάρχει, ο Γέννης έχει ομάδα επισκεπτών επίσης ε, παρούσα εδώ, οπότε έχει δικαίωμα να μιλήσει περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και λαμβάνετε υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα. Κυρία Επίτροπε, οι συζητήσεις ε, συχνά στρέφονται προς το παρελθόν και κοιτάμε το τι συνέβη. Πρέπει όμως να δούμε και τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Συμφωνώ μαζί σας, Επίτροπε πρέπει με βιώσιμο τρόπο να δούμε το πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές, να εξετάσουμε το θέμα της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της ε, ε, βιομηχανίας. Είπατε κι εσείς ότι πρέπει να κουνηθεί η βιομηχανία, να κινηθεί στο θέμα της κινητικότητας και είπατε ότι στο θέμα των μπαταριών δεν έχουμε μεγάλη ε, πρόοδο. Πολιτική σημαίνει εξέταση της πραγματικότητας ο Υπουργό Οικονομικών τη Γερμανία είναι έτοιμο να δώσει 1,7 δισεκατομμύρια για μπαταρίε. Έτσι είπε. Τελικά δεν θα τα δώσει. Χρειάζεται όμω να γίνουν σωστοί οικονομικοί υπολογισμοί. Συμφωνήσαμε με ανώτατα όρια για, για ε, αυτοκίνητα και για τα φορτηγά. για τα αυτοκίνητα συζητάμε μόνο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι και αυτό με βρίσκει επικριτικό. Λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε μια ουδετερότητα τεχνολογική, πρέπει να δούμε εναλλακτικά κάψιμα, ε, εναλλακτικές λύσεις ενεργειακές. Θέλετε καινοτομία, είσαστε η Επίτροπος υπεύθυνη για θέματα βιομηχανίας και πρέπει να το κάνετε αυτό διότι αν ανταλλάξουμε βρώμικο ντίζελ για μια μορφή ενέργειας ακόμα πιο βρώμικη, όλοι θα χάσουμε το παιχνίδι. Έχετε κάτι ε, καθοδόν. Σε αυτά που είπατε είσαστε κάπως επιφυλακτικοί. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια ημερομηνία συγκεκριμένη, να τη σημειώσω και να δω κατά πόσο σας συμμορφωθείτε με την υπόσχεσή σας. Έχουμε δύο ομιλητές των σοσιαλιστών στον κατάλογο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από 1,5 λεπτό. Ορίστε. Ευχαριστώ. Θέλω να ξέρω αν κατάλαβα καλά. Είχαμε την Επιτροπή, την ΕΜΙ, την ερευνητική που είπε ότι είναι κακό η Τεχνική Επιτροπή για, τα, για τις κινητήρες οχημάτων να τροποποιήσει πολιτική απόφαση για τους παράγοντες συμμόρφωσης. Είχατε την απόφαση του ΔΕΚ. Οι πόλεις θέλουν περισσότερες φιλοδοξίες, φιλόδοξους στόχους και είπε το ΔΕΚ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να τροποποιήσει ε, τους κανόνες εκπομπής για τις νέες δοκιμές υπό συνθήκες οδήγησης. Εσείς στις παρατηρήσεις είπατε ότι το δικαστήριο δεν επετέθη κατά των παραγόντων συντελεστών συμμόρφωσης. Ο συντελεστής συμμόρφωσης δεν είναι κάτι νόμιμο. Κουνάτε το κεφάλι σας. Πώς ερμηνεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει το ΔΕΚ, δεν μπορούσε να τροποποιήσει το, τα όρια εκπομπών Euro 6 για τις δοκιμές πραγματική οδήγηση. Τώρα, αν εφεσιβάλλετε την απόφαση εν ώψη νέας δεν υποβάλλεται μόνο μία νέα κατεξουσδότηση πράξη για να απαλλαγείτε από την παλιά ε, κατεξουσδότηση πράξη που το 10 έκρινε παράνομη. Αντί να κάνετε να ακολουθήσετε ταχεία και απλή διαδικασία, τι προτείνετε να κάνετε. Νέα νομοθεσία, συναπόφαση, που θα χρειαστεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με την επιφύλαξη του αποτελέσματος της έφεσης. Άρα τελικά ε, θα αποδυναμωθούν οι στόχοι μέσω αυτής της διαδικασίας και αυτής της νομοθεσίας. Αλλιώς δεν έχει αυτή η προσέγγιση σκοπό. Μετά λέτε ότι μειώνουμε τους στόχους που σχετίζονται με το συντελεστή συμμόρφωση, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα αν γίνει αυτό και παρετούμεθα τη έφεση. Αυτό είναι πολύ κακό που κάνετε. Η κατεξοδότηση πράξη είναι η απλούστερη λύση είναι η σωστή λύση στο πνεύμα της απόφασης του ΔΕΚ. Δεύτερον, πραγματικά πιστεύετε ότι το Κοινοβούλιο θα θεσπίσει νομοθεσία για να μειώσει τους στόχους εκπομπών, δοθέντος αυτών που γνωρίζουμε και αυτών που είπαμε για το θέμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά ελπίζω εγώ να μην έχω καταλάβει, να κάνω λάθος. Διότι αυτά που είπατε μου φαίνονται άκρος παράξενα. Ευχαριστώ. ECR. Μάρκ, ξανά για ένα λεπτό. Α. Δεύτερη ερώτηση των σοσιαλιστών. Μπονφουά. Για ένα μισή λεπτό. Κυρία Μπονφουά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την εδώ παρουσία σας. Και εγώ θα επανέλθω σε αυτή την απόφαση του 10 του Δεκεμβρίου. Διότι η υπόθεση ήταν προσφυγή των Παρισίων, των Βρυξελών, της Μαδρίτης. Προσέφυγαν οι πόλεις, διότι αντιμετώπιζαν πολύ μεγάλη ρήπανση και ανησυχούσαν πάρα πολύ από τον ε, συντελεστή συμμόρφωση στη πραγματικότητα ε, δεν εφαρμόστηκε. Να βάλουμε ένα ακόμα κάτι δεν σημαίνει ότι έχουμε ένα πρότυπο συμμόρφωση και σεβασμού και τα αποτελέσματα είναι ότι κάτι και αυτών των πόλεων πλήττονται από αυτή την ψηλή, τη μεγάλη ρήπανση. Λέτε ότι εταιρείε και η κοινωνία αλλάζει επίσης αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί εμεί, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν καταλαβαίνει η κοινωνία, γιατί δεν σεβόμαστε τι προδιαγραφέ που εμεί καθορίσαμε μέσω των συντελεστών συμμόρφωση. Ε, δεν θα πρέπει να περιμένουν τώρα για νέο δικό χάρτη, για νέε συζητήσει. Ο κόσμο τι χρειάζεται. Χρειάζεται αποφάσει που λαμβάνονται και που γίνονται πραγματικά σεβαστέ και γίνονται σεβαστέ από όλου. Ε, προχωράτε, αλλά όχι αρκετά γρήγορα έναντι της καταστάσεως που αφορά την ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη που δεν βελτιώνεται και θα πρέπει να ληφθούν με υπεύθυνο τρόπο μέτρα. Μία ερώτηση λοιπόν σχετικά με την Τεχνική Επιτροπή για τα οχήματα. Κάτι που το συζητήσαμε στην Επιτροπή Ερεύνας και εκεί είχαμε καταγγείλει την έλλειψη διαφάνειας. Πού βρίσκονται οι εργασίες για να προχωρήσουμε πως, ε, μια, για προδιαγραφές Euro 7 διότι είναι δρόμος χωρίς επιστροφή αυτός, το χρειαζόμαστε αυτό. Μήπως όπως και με το παράγοντα συμμόρφωση σε ένα δεν θα προχωρήσουμε και εδώ. Είπατε ότι σε τέσσερα χρόνια τελικά θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο στόχο. Παρόλο που το θέμα εδώ και δύο χρόνια έχει τεθεί επιτάπητος. Πρέπει να προχωράτε πιο γρήγορα, κύριε Επίτροπε. Ε, ευχαριστώ. Άλτε. Ο κ. Γκερμπράντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Φοβούμαι ότι η Επίτροπος δεν με έπεισε απόλυτα με τι απαντήσει τη στον πρώτο γύρο. Αν η απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούσε το σώμα, το κολέγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει στι τάξει αυτή τη θέση τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε στην απάντησή σα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε κάποιε ερωτήσει. Και αυτό διότι αυτά τα θέματα εμπίπτουν στα προνόμια του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν ανήκει σε αυτή τη συλλογική, εντάσσεται τη συλλογική απάντηση, τότε και το προνόμιο του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσεται στο κολέγιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται στα πλαίσια αυτή τη κοινή απάντηση τη Επιτροπή στο σύνολό τη. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί αυτά τα θέματα που εμπίπτουν στα προνόμια και δικαιώματα του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτά δεν συμπεριλήφθησαν στην απάντηση και αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν το κατανοώ. Δεύτερον, να απαλλαγούμε από από τα οχήματα αυτά τα πατηλάου του ΣΥΠΗΝ που ακόμα κυκλοφορούν. Είναι και αυτό το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελεκτικό συνέδριο. Πρέπει να ε, επιληθεί. Τώρα αναφερθήκατε για κάποια συνάντηση το Μάρτιο που δεν είναι πολιτική φύση, περισσότερο τεχνική. Αυτό δεν είναι κάτι που αρκεί. Αυτή η συνάντηση δεν αρκεί. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ηγηθεί. Και αν χρειαστεί και σε επίπεδο Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν έχει χρόνο να αντιμετωπίσει το χρόνο τον, τον θερινό και το χειμερινό, σίγουρα έχει και χρόνο να αντιμετωπίσει και ένα θέμα που προβληματίζει 500 εκατομμύρια ανθρώπου και επηρεάζει την προσωπική του υγεία. Γιατί δεν εμπλέκεται προσωπικά ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γιατί οργανώνει με τεράστια σύνοδο κορυφή για την απαλλαγή από τα βρώμικα αντιζελοκίνητα οχήματα, να εξυγχρονιστεί και το λογισμικό και ο εξοπλισμό ομοιόμορφα στην Ευρώπη και όχι μόνο βάσει των θετικών ιδεών ε, διαφόρων υπουργών ε, κρατών μελών. Νομίζω ότι οι πολίτες μας αξίζουν πολλά περισσότερα από αυτά που μας ε, δίνεται τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ίσως να, να πάρει και μία ώρα το χειμερινό χρόνο, τη χειμερινή ώρα για να το διοργανώσει. Η FDD ήταν στον κατάλογο για το δεύτερο γύρο. Δεν ήταν μάλλον στο, στο κατάλογο. Είμαστε καλοί. Όμως η Λεωνόρα έχει μια ερώτηση και της επιτρέπουμε τη Λεωνόρας να την υποβάλει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ νέου, μια ερώτηση εντάχει για το θέμα αυτών των ανακλήσεων και των αποσύσεων. Κυρίως για τη χώρα μου, για την Ιταλία, οι ε, ανακλήσεις και όσον αφορά και το Volkswagen, τη Volkswagen και άλλες εταιρείε έχουμε στοιχεία τα οποία δεν φαίνονται να είναι σύγχρονα επικαιροποιημένα. Χρονολογούνται από τον Ιανουάριο του 2018. Μπορείτε να μας δώσετε πιο σύγχρονα στοιχεία όσον αφορά τις ανακλήσεις οχημάτων. Ε, μετά μία ερώτηση άλλη. Πώς βλέπετε τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Volkswagen και της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε την έκθεση της Όλαφ για 400, εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η Volkswagen πήρε από το 2000 2014 που δεν χρησιμοποίησε για να προωθήσει καθαρές τεχνολογίες αλλά για να, βρει, να εφεύρει αυτές τις ε, συσκευές παράκαμψης. Υπήρξε λοιπόν συμφωνία ε, στις 20 Δεκεμβρίου που συνήθει μεταξύ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Volkswagen για 10 εκατομμύρια ευρώ που δίνονται για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. έχετε κάποια σχόλια όσον αφορά αυτή τη συμφωνία, αυτή τη συμφωνία. Πολύ γρήγορη η ερώτηση αυτή. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο δεύτερο γύρο. Μπορούμε να επιστρέψουμε στην ε, Επίτροπο να δώσει απαντήσει. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω εκ νέου με την απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ είμαι πολύ σίγουρη για αυτά που λέω. Η απόφαση αφορούσε τη διαδικασία, ουχή το περιεχόμενο. Αυτό είναι, το νομικό, είναι νομικό πρόβλημα και έχει πρόβλημα επί της ουσίας, επί του περιεχομένου, του συντελεστού συμμόρφωσης. Το Κοινοβούλιο το παρόν και το μελλοντικό θα συζητήσει την νέα πρόταση για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι η κατεξοδότηση πράξη δεν είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος. Γι' αυτό πρέπει να προτείνουμε νέα πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Και γι' αυτό έδωσα την πρώτερη εξήγησή μου. Μπορώ να σας δώσω κάποια ενημέρωση νομικού περιεχομένου από αυτού. Αλλά είμαι 100% σίγουρη ότι η απόφαση ήταν όχι η κατεξοδότηση πράξη, αλλά νέα διαδικασία μέσω συναπόφασης. Και δεσμεύομαι ότι θα σας δώσουμε νέα πρόταση σε μία εβδομάδα. Ούτε εβδομάδες. Τέλος πάντων, σύντομα, αν δεν είναι μία εβδομάδα, πολύ σύντομα. Θα έχουμε την ίδια βάση αφορά τη διαδικασία και όχι το περιεχόμενο. Είμαι απόλυτα βέβαιη γι' αυτό. Για την τεχνολογική ουδετερότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την πλευρά μου προσωπικά πρέπει να πω ότι πάντα μιλάμε για οχήματα με μηδενικές εκπομπές όχι μόνο ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα οποιαδήποτε οχήματα να μην εκπέμπουν Θέλουμε οχήματα μηδενικών εκπομπών. Υβριδικά, ηλεκτροκίνητα, αυτόματα, στρατηγική προσέγγιση ευρωπαϊκή. Και για αυτό το πλαίσιο επιτρέψαμε πολλές κρατικές επιδοτήσεις. Αυτό επεξεργαζόμεθα. Οι ανταγωνιστές μας στον υπόλοιπο κόσμο κινούνται τάχιστα. Ε, Κυρίως όσον αφορά τα ηλεκτριοκίνητα αυτοκίνητα. Και όπως σας είπα, αν η βιομηχανία μας δεν κινηθεί πολύ ταχύτερα από ό,τι μέχρι τώρα, τότε θα έχουμε πρόβλημα με θέσεις εργασίας και με ανταγωνιστικότητα και την παρουσία του τομέα μας αυτού του ευρωπαϊκού στον κόσμο. Για τις ε, ανακλήσεις. Για τις ανακλήσεις στην Ιταλία τέθη μια ερώτηση. Όπως προανέφερα. Πριν από ένα χρόνο είχαμε νέα στο σελίδα που δημιουργήσαμε. Επικαιροποιείται καθημερινά και έχουμε ενημερωμένα στοιχεία από κάθε κράτος μέλος όσον αφορά τις ανακλήσεις. Δεν ξέρω τα στοιχεία για την Ιταλία, μπορείτε να τα βρείτε εύκολα. Μπορούμε να σας δώσουμε τις δέουσες πληροφορίες για το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη Volkswagen. Έχουμε ελέγξει την περίπτωση, διεξοδικά δεν βρήκαμε κάτι παράτυπο. Δεν έχουμε βάση να κινηθούμε, να αντιδράσουμε. Αυτά νομίζω. Α, γύρω πέντε. Πέντε, τι πέντε, τι λέω. Επτά μου δίνουν εδώ, βλέπω, ε, πέντε διαβάζω εγώ. Τι να κάνω. Λοιπόν, στα πλαίσια συναπόφαση. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί και θα ενημερώνεται πλήρω. δεόντως, δεν θα είναι έργο τεχνικής επιτροπής. Ξεκίνησε πέρσι η εργασία. Και τώρα εξετάζουμε το πεδίο εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Ίσως και φέτος, κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, ίσως να υπάρξει κάποια πρόταση που θα επεξεργαστεί το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της νέας του σύνθεσης. Αυτά, ευχαριστώ. Α, αν κάτι ξέχασα, κάποια ερώτηση, θα προσπαθήσω να σας δώσω απάντηση γραπτός να σας επιστήσω την προσοχή σε κάτι άλλο. Τα ξέρετε όλα απ' έξω και ανακατοτά, αλλά να, αυτό είναι το φυλάδιό μας. Είναι πολύ ωραίος τρόπος παρουσίασης των συλλογικών μας επιτεγμάτων τα τελευταία 3,5 χρόνια. Κάπου εκεί το έχουμε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Η κυρία Βαν έχει μια ερώτηση. Ναι, ναι, μια παράκληση, όχι τίποτα επί του περιεχομένου. Να σας παρακαλέσω λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτά που σκέφτονται οι ευρωβουλευτές ε, σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου και σχετικά με αυτά που μας λέτε, ε, να συνδυαστεί η μεθοδολογία με το περιεχόμενο. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ενημέρωση από εσάς για το πώς ερμηνεύετε εσείς την απόφαση του δικαστηρίου και ε, τι θα περιλαμβάνει η πρόταση αλλαγής που θα υποβάλλετε. Διότι μην ξεχνάτε, αν καταθέσετε μία νέα πρόταση οδηγίας με την ε, συμμόρφωση ως παράγοντα, ε, τότε δεν θα έχετε τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Ίσως είναι το τελευταίο που μπορούμε να κάνουμε πριν τις ευρωεκλογέ, ε, αλλά θα μπορούσατε να συντάξετε ένα ανεπίσημο έγγραφο, ένα non-paper την άλλη εβδομάδα, ας πούμε. Θα μας βοηθούσε πάρα πολύ ή τις επόμενες εβδομάδες. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο είναι χρήσιμο, διότι έτσι θα μπορούμε να προετοιμαστούμε για την επόμενη θητεία, γιατί θα αναγκαστούμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα τότε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στις επόμενες τρεις μέρες θα σας ε, διαβάσουμε την νομική ανάλυση για να την διαβάσετε. Και νομίζω ότι ότι στην τελευταία συνεδρία στην Επιτροπή ΕΜΗΣ ε, θα έχω τη δυνατότητα να συναντηθώ με εσάς για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ελάχιστο χρόνο που διαθέτουμε για να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε τη μετάβαση έτσι ώστε η επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, το επόμενο κοινοβούλιο να ε, πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πίτροπε. είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία, διότι όταν τα πράγματα μένουν στα χέρια των ε, δικηγόρων, τότε η κατεύθυνση που παίρνουν τα πράγματα είναι διαφορετική από αυτή που περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πίτροπε. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά που σας βλέπουμε, αλλά θα δούμε. Τώρα θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Okay, ready to go. Αν είστε έτοιμοι, τότε μπορούμε να περάσουμε στο ε, επόμενο θέμα για τις, ε, τον προσδιορισμό των πρώτων υλών που ενέχουν υψηλό κίνδυνο έμεση αλλαγής της χρήσης της γη. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί για περίπου 1,5 χρόνο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φανιστή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω το σχέδιο πράξης κατεξουσιοδότησης για ε, τα ε, καύσιμα που έχουν υψηλό κίνδυνο έμεσης αλλαγής χρήσης της γης. Παρουσίασα την πρόταση αυτή στην Επιτροπή Ήτρα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα την παρουσιάσω και εσάς, σε εσά σήμερα το απόγευμα. Το σχέδιο πράξη κατά εξουσιοδότηση λοιπόν έχει ήδη δημοσιευθεί για να διανύσουμε την ε, περίοδο τεσσάρων εβδομάδων κατά την οποία θα λάβουμε τα σχόλιά σας και τις εντυπώσεις σας. Θα σας ε, παρουσιάσω την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι να φτάσει στην ε, μορφή που έχετε σήμερα, αλλά θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια αναδρομή στο πλαίσιο και στο παρελθόν το οποίο την οδήγησε, οδήγησε στην ε, πρόταση αυτή. Πρέπει να δούμε λοιπόν τη γενικότερη εικόνα, δηλαδή την ε, οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αναθεώρησή της την αναδιατύπωση μάλλον που εγκρίθηκε πέρυσι. Η νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως γνωρίζετε, έχει ως κύριο σκοπό να προωθήσει την ανανεώσιμη ενέργεια όλων των μορφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων και των ε, ε, ε, και συμπεριλαμβανομένες της ανανεώσιμης ενέργειας προέρχεται από βιοκαύσιμα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό εντοπίσαμε τις κύριες προϋποθέσεις για να εντοπίσουμε τα βιοκαύσιμα με υψηλό κίνδυνο έμεσης αλλαγής χρήσης της γης. Εν συντομία, στην οδηγία υπάρχει ένα όριο για το πόσα βιοκαύσιμα μπορούν να παραχθούν και να προσμετρηθούν στον στόχο του 2020. Για το 2020 λοιπόν το ανώτατο όριο είναι 7% όμως ε, το κάθε κράτος μέλος μπορεί να θέσει τα δικά του όρια. Αυτό είναι συνέχεια της προηγούμενης ε, προσέγγισης που είχαμε υιοθετήσει για την έμεση αλλαγή χρήση της ε, γης, στην οδηγία ILUC δηλαδή του 2015. σε ό,τι αφορά τα νέα κριτήρια. Δηλαδή, με τα βιοκαύσιμα υψηλού κινδύνου πρόκειται να παγώσει η ε, συνεισφορά των ε, καυσίμων αυτών ε, προς τον στόχο για το 2021 μέχρι το 2023. Το 2019 θα παγώσει το, το ποσοστό αυτό στα, σε επίπεδο κρατών μελών και το 2023 θα γίνει μια σταδιακή κατάργηση αυτού του είδους βιοκαυσίμων μέχρι το 2030 έτσι ώστε να φτάσουμε στο μηδέν. Επιπροσθέτως, υπάρχει και μια εξαίρεση για τα βιοκαύσιμα χαμηλού κινδύνου έμεσης αλλαγής χρήσης της γης. Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σαφέστατα στην οδηγία ότι μπορεί να συνεχίσει να παράγεται από πρόσθετες πρώτες που προκύπτουν από, ε, σοδιέ, από αυξημένες ε, σοδιές, που δεν επηρεάζουν καθόλου δηλαδή την χρήση της ε, γης. Είναι σύμφωνα με το σκεπτικό της οδηγίας δηλαδή. Δηλαδή, αυτό που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να οριστούν οι προϋποθέσεις για την παραγωγή την, ε, και την ε, επέκταση της καλλιέργειας αυτών των βιοκαυσίμων και αυτό έγινε τώρα, γι' αυτό διηγηθήκαμε στην ε, δημοσίευση του σχεδίου πράξης κατά εξουσιοδότηση. Και η έκθεση που έχουμε ετοιμάσει είναι αποτέλεσμα της ε, διαβούλευσης με τους εμπειρογνώμονες. Αυτό δηλαδή που προτείνουμε δεν είναι μια νέα πολιτική, είναι τα κριτήρια της προσέγγισης, πάνω στα οποία κριτήρια έχουν ήδη ε, αποφασίσει οι συνομοθέτες και τα έχουν εγκρίνει. Το σχέδιο είναι λίγο πολύ απλό. Πρώτα, τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται σε καύσιμα υψηλού και χαμηλού κινδύνου, σε εκείνα που, συγκε... που πληρούν ε, συγκεντρωτικά τις προϋποθέσεις, δηλαδή ελάχιστη, μάλλον επέκταση στο ελάχιστο της ε, επιφάνειας καλλιέργειας, ως 100.000 εκτάρια ανά έτος και το πιο σημαντικό προτείνουμε τα καύσιμα αυτά να καλλιεργούνται όχι πάνω από το, ε, σε, σε επιφάνεια όχι πάνω από το 10% εδαφών τα οποία έχουν υψηλό, υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Νομίζω πως αυτά τα κριτήρια συμπεριλαμβάνουν όσα έχουν ζητήσει από εμάς οι νομοθέτες. Γιατί τα βιοκαύσιμα αυτά έχουν αμέσω επιπτώσεις σε εδάφη με υψηλή συγκεντρώση άνθρακα και τα βιοκαύσιμα που θα προωθούνται με την νέα οδηγία θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Και δεν θα κινδυνεύει να χαθεί η βιοπικιλότητα. Αυτά προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε. Τώρα, στοιχεία για τα επίπεδα της επέκταση αυτή. Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στην έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε μαζί με το σχέδιο πρότασης κατά εξουσιοδότηση. Και σύμφωνα με την οδηγία, τα είδη καυσίμων Υπάρχουν συγκεκριμένα μάλλον είδη καυσίμων που δεν ε, θα καλλιεργούνται μετά το 2023 και ε, θα σταματήσουν τελείως μέχρι το 2030. Τώρα, τα βιοκαύσιμα χαμηλού κινδύνου αλλαγής χρήσης της γης. Υπάρχουν και εδώ ορισμένα κριτήρια. Συγκεντρωτικά υπάρχουν τα κριτήρια για τη βιωσιμότητα που περιέχει οδηγία Έπειτα υπάρχουν τα βιοκαύσιμα τα οποία προέρχονται από πρόσθετες πρώτες ύλες που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα της ε, καλλιεργής γης που ήδη καλλιεργείται, αλλά και γης η οποία μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιούταν, ήταν εγκαταλειμμένη ή καλλιέργητη. Φυσικά θα υπάρχει ενδελεχής έλεγχος της όλης διαδικασίας. Για να φτάσει η αύξηση της παραγωγικότητας πέρα από τα όρια τα οποία περιγράφονται στην οδηγία, υπάρχουν ορισμένα πρόσθετα κριτήρια για τη δημιουργία ε, συστημάτων καθαριότητας και η καλλιέργεια αυτή θα περιορίζεται σε ένα ανώτατο διάστημα 10 ετών, το οποίο νομίζουμε πως είναι αρκετά λογικό. Τέλος, υπάρχουν ορισμένα πλουστευμένα κριτήρια σε ορισμένες ε, ξεκάθαρες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ακαλλιέργητη γη, υποβαθμισμένη γη ή πολύ μικρές ε, μονάδες. Θεωρούμε λοιπόν συμπερασματικά ότι η προσέγγιση μας είναι αρκετά εξισορροπημένη, στηρίζεται από επιστημονικά στοιχεία και πάνω απ' όλα είναι μια πρόταση η οποία συμμορφώνεται απόλυτα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βέβαια, κατανοούμε ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, γι' αυτό προβλέπεται προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και να είστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί αδιαλείπτως τις εξελίξεις και μέχρι το 2021, δηλαδή σύντομα, θα γίνει αναθεώρηση και των ε, πιο πρόσφατων επιστημονικών ε, στοιχείων, αλλά και της προσέγγισης που έχουμε υιοθετήσει. Όπως σας είπα, έχει δημοσιευθεί το σχέδιο της πράξης κατά εξουσιοδότηση. Βρισκόμαστε στη διαδικασία της ε, δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τις 8 Μαρτίου. Μόλις, ολοκλη... Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να, να εγκρίνουμε την ε, πράξη το συντομότερο και να ξεκινήσει επίσημη διαδικασία στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Επίσης, πρωτού λήξει η περίοδος ε, διαβούλευσης, θα συσταθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, θα συνεδριάσει στις 5 Μαρτίου. Αυτά από εμά, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά θα ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τυχόν σχόλια ή ερωτήσει που μπορείτε να έχετε σε αυτό το στάδιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στίν. Μπορούμε τώρα λοιπόν να περάσουμε στου σκιώδει, που είναι 1,5 σκιώδη ουσιαστικά στην αίθουσα και στον εισηγητή. Ο κύριο Άκουτ, παρακαλώ, πρώτος. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και εγώ, Χάνς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας εξήγησε αυτή την κατεξουδιώτηση πράξη που τέθη σε ψηφοφορία μετά από δικό μας απερίφραστο αίτημα και ξέρετε τι συμβαίνει. Θέλουμε εμείς το φινικέλο να το ε, απογορεύσουμε, ε, να μην χρησιμοποιείται ως ε, βιώσιμη πηγή για τις ΑΕΠ και είπαμε Κομισιόν να μας καταθέσει τα κριτήρια. 1η Φεβρουαρίου η τελική προθεσμία. Λίγο καθυστερημένη λοιπόν, αλλά εντάξει. Και ξέρω πως κάνατε και κάποιες διαπραγματεύσεις με την Digitrade. Trade. Καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν απαραίτητο. Κάνα δύο ερωτήσεις. Μπορούμε να επαναλάβουμε τις επικρίσεις τις οποίες ακούστηκαν χτες στην Ήτρε. Και θα είμαι σαφής. Το ΕΛΚ, το, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι, οι πράσινοι και οι γκου ήταν όλοι πολύ επικριτικοί. Οπότε καλό θα ήταν να ακούσουμε λίγο τι είδου αλλαγέ προβλέπετε εσεί, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαβούλευση και πρέπει να σα πω πω θα ακούσετε πάρα πολλέ επικρίσει και από τη διαβούλευση. Πείτε μου λοιπόν, θα αλλάξετε κάτι ή απλώ εδώ το κάνουμε για να φαίνεται. Και επίση, τι είδου αλλαγέ. Και να σα βοηθήσω πρώτα απ' όλα, το κατόφλι του 10% από πού προέρχεται, πώς αιτιολογείται. Γιατί αν δείτε το παράρτημα θα δείτε το φινικέλαιο εμπίπτει στο phase out, αλλά όχι η σόγια. Παρόλο που και η σόγια έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις αυτό, ελπίζω να μην σχετίζεται με το Γιόνκερ που τον Ιούλιο πέρσι πήγε στις Ηνωμένε Πολιτείες και θα ήθελα να πείτε αν το κατόφλι το 10% έχει επιλεγεί για να είναι η σόγια κάτω από το κατόφλι και να είμαστε ασφαλείς εκεί με τη σόγια και όχι το φινικέλαιο. Γιατί βέβαια όπως ήταν πολύ δύσκολο να αποκλείσετε το φινικέλαιο, το είχαμε δει αυτό από την αρχή. Αν όμως τελικά γνωρίσετε πως το φινικέλαιο αποτελεί πραγματικά αρνητικό σημείο για την ε, αποψήλωση των δασών και θέλετε να συμφωνήσετε μαζί μας ότι δεν είναι βιώσιμο, τότε ε, θα πρέπει να δούμε ε, εάν ε, το προσπαθείτε να το ξαναεντάξετε μέσω του Low Island Group. Δηλαδή, γεές που δεν είναι σε χρήση. Τι σημαίνει αυτό, γές που δεν είναι σε χρήση γεωργική, λέει ο ορισμός. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει, ή λοιπόν γεωργική χρήση ή καμία χρήση. Γνωρίζει η Επιτροπή πώς μπορεί η γη να χρειαστεί για παράδειγμα, για να μένει ο κόσμος επάνω στη γη. Γιατί λοιπόν η μη χρησιμοποιημένη γη είναι τόσο περιοριστικά ορισμένη, ώστε να υπάρχει τέτοιο τεράστιο απόθεμα μη χρησιμοποιημένων γεών. Πείτε μου λοιπόν στον ορισμό θα αλλάξετε κάτι. Και επίσης για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή, αν είστε μικρή εκμετάλλευση είστε εντάξει. Μα στη Μαλαισία για παράδειγμα, όλες οι μικρές εκμεταλλεύσεις εκεί δουλεύουν για μεγάλες ε, πολυεθνικές. Αλλά τους λέμε μικροεκμεταλλεύσεις γιατί στον ορισμό αυτό λέει θα πρέπει κανείς ή να ενοικιάζει γη ή να μισθώνει γη ή να έχει την κατοχή του γη. Τι θα αλλάξει αυτό στη Μαλουσία που εκμισθώνουν γες από τις μεγάλες εταιρείε οι, αγρότες και αυτό τους απαλλάσσει. Δηλαδή, είναι πάντα σε συμμόρφωση και μπορούν να συνεχίσουν όπως σήμερα. Τι σημαίνει αυτό για τις τρέχουσες πρακτικές, τι θα αλλάξει και τέλος πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά. Πιστοποίηση λέει όπου θα αποδεικνύουν ότι θα έχουν επιπλέον αποδόσεις στις οδιές τους. Τι σημαίνει αυτό. Σε κάποιες χώρες θα πούνε εμείς θα τους δώσουμε την πιστοποίηση και μετά θα συνεχίσουν τα πράγματα όσοι έχουν. Οπότε παριστάνετε ότι κάνετε αυτό το phase out με τις ε, εξαιρέσεις ε, για το χαμηλό κίνδυνο, ουσιαστικά εξαιρείται όποιον εργάζεται σήμερα. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει κάτι business as usual. Αλλά δεν ήταν αυτή η πρόθεση της κατεξοδότηση πράξης, οπότε θα ήθελα να πείτε ακριβώς για το 10% και για τις μη χρησιμοποιημένες γέες και για τις μικρές εκμεταλλεύσεις και το πώς θα εφαρμόσουμε το τι θα συμβούν. Γιατί μετά η Ιταλία και η Ισπανία θα πούνε εντάξει πιστοποιημένοι είναι, συνεχίζουμε όπως πριν. Και θα δούμε εμείς ε, την άποψη ε, ψήλωση των δασών που θα συμβαίνει για τα βιοκαύσιμα και αυτό είναι αυτό που θέλαμε να παρεμποδίσουμε και νομίζω ότι με τις δικές σας εξαιρέσεις δεν θα το καταφέρουμε. Η κυρία Πετήρ, παρακαλώ. Όχι. Αντικαταστάτηση, κυρία Ντελέ. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, η συνάδελφος δεν είναι εδώ. Θα διαβάσω εκ μέρους της όμως το κείμενο το οποίο ήθελε να παρουσιάσει σε ανησυχώ από το κείμενο που προτείνεται για το σχέδιο της κατεξοδότησης πράξης, γιατί αφεμάσει το αρχικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι η μείωση αυτών των βιοκαυσίμων που δεν είναι βιώσιμα, μειώνοντας την ε, ε αποψήλωση των δασών. Αυτό δεν συμπίπτει καθόλου με τους στόχους μας έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Γιατί έχουμε αυτές τις εξαιρέσεις για το ε, χαμηλό κίνδυνο και είναι ε, πολύ ε, πάρα πολύ δύσκολο να δούμε ποιες, πώς θα επηρεάσει αυτό την εμπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, μικρές ποσότητες ή μεγάλες ποσότητες φινικηλαίου μπορούν μέσω αυτής της εξαίρεσης να μπαίνουν μήπως θα πρέπει να δούμε αυτούς τους περιορισμούς του άρθρου 5, από τους οποίους εξαιρεί τους μικροκαλλιεργητές ξανά. Για την ανάλυση κινδύνου δεν λάβαμε στοιχεία παρόλη την πολιτική, οικονομική και οικολογική σημασία αυτού του φακέλου και δεδομένου ότι η πολιτική μας είναι να κάνουμε καλύτερη νομοθεσία θεωρούμε πως αυτή η κατοξιοδότηση πράξη είναι προβληματική. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα Κανέσουνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συνεχίσω τα όσα είπε ο συνάδελφος, γιατί πιστεύω ότι ήταν πραγματικά πολύ γλαφυρός και θέσε πολλές ερωτήσεις. Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή ε, που εγκρίναμε το πρώτο μήνυμα για το τι ακριβώς αποτελεί φινικέλαιο, καταλήξαμε στο εξή. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια στα κείμενά μας λέγαμε πως το φινικέλαιο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ότι δεν μπορούμε να λέμε απλώς το φινικέλαιο έτσι απλά. Εσείς λέτε ε, φινικέλαιο, ε, απώλεια δασών, ε, τεράστιο πρόβλημα, ε, και άρα λοιπόν τα βιοκαύσιμα που έχουν φινικέλο δεν μπορούν να θεωρηθούν πως ε, συμβάλλουν στο βιώσιμο περιβάλλον. Και στο έγγραφό σας σήμερα ξαφνικά δηλώνεται ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή εμείς σας ζητάμε ε, να κάνετε το αντίθετο. Δεν νομίζω ότι αυτό δείχνει σεβασμό προς το Κοινοβούλιο, γιατί με το φινικέλο σε αυτό το έγγραφο κάνετε κάτι εξιοπερίεργο. Και έχω μόνο μία ε, ε, επιπλέον ερώτηση σε σχέση με τον συνάδελφο. Και η οποία είναι η εξή. Πόσο συχνά έχετε συναντηθεί με τους λομπίστες του Φινικελαίου από τη Μαλισία και την Ινδονησία πριν παρουσιάσετε αυτά. Και πρόκειται εδώ για κάποιο είδους ε, ανταλλαγή με κάποιο όφελος που θα σας προσφέρουν η Μαλαισία και η Ινδονησία. Γιατί λέτε πως έχουν όλα και επίσης εξαιρείται τις μικρές φυτίες μέχρι 5 εκτάρια. 99% λοιπόν από αυτές δεν συμμορφώνονται με τα ε, κριτήρια και τις απαιτήσει. Και αυτό εις βάρος του πληθυσμού της Ινδονησίας και της Μαλαισίας. Και δεν εξηγήσατε καθόλου πώς οι φυτές αυτές θα ελέγχονται. Και πείτε μου, συμμορφώνονται με όλα τα δικά μας περιβαντολογικά ε, κριτήρια, με το σεβασμό των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων. Γιατί αυτό που περιγράφεται είναι κάποιο σενάριο που προέρχεται από άλλη γενική διεύθυνση, αλλά εμείς περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Ένα έγγραφο το οποίο θα ευθυγραμμίζεται με αυτά τα οποία ζητήσαμε εμείς εδώ και χρόνια, εδώ και τρία χρόνια ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μην περιμένετε πως εμείς αυτό το έγγραφο θα μπορέσουμε να το δεχτούμε και ότι θα πούμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε στη μάχη κατά της αποψηλωσής των δασών. Γιατί τα πρακτικά βήματα που θα ακολουθήσουν, ε, σύμφωνα με αυτό, δεν θα μας βοηθήσουν καθόλου. Και ξέρετε τι λέμε στο Jurassic Park, η ζωή βρίσκει τον τρόπο πάντα, αλλά Νομίζω ότι τελικά τον τρόπο που βρήκε, ε, αυτός που βρήκε κάτι σε αυτή την περίπτωση ήταν οι λομπίστες που βρήκαν την πόρτα του γραφείου σας και με, λυπάμαι πάρα πολύ που τα λέω έτσι. Θα το επαναλάβω λοιπόν αυτό, αν χρειαστεί. Γιατί, γιατί η σόγια δεν είναι ο κομμάτι στον κατάλογο ε, με τους ε, υψηλού κινδύνου. Υπάρχει απάντηση. Η κυρία Ντελέη θα μιλήσει εξ ονόματής της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, θα μιλήσω εν ονόματί μου. Μπορούμε να συμφωνήσουμε και να στηρίξουμε προς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την του του φινικελαίου. Το να βάλουμε εξαιρεσει που προτείνει νομίζω ότι αντιστοιχεί σε, στο να αυτοκοροϊδευόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μία εξαίρεση για τους μικρούς παραγωγούς. Τι εννοούμε με αυτό, ποιος είναι ο μικρός παραγωγός. Καθένας ξέρει λοιπόν ότι οι μικρές ταγόνες κάνουν το μεγάλο ποτάμι. Αυτή η εξαίρεση για τους μικρούς παραγωγούς νομίζω ότι είναι κάτι αδικαιολόγητο. Και προφανώς θα οδηγήσει σε διπλασίαση της εξαγωγής του φινικελαίου που θεωρήσαμε ότι είναι κάτι μη εγκρίσιμο στην ε, Ευρώπη. Το θέμα της προσθετικότητας. Κανένα κριτήριο αξιολόγηση δεν προτείνεται και αφήνουμε στους συμμετέχοντες την εξακρίβωση του τι σημαίνει αυτό, να το κάνουν οι ίδιοι. Ε, Δη, δηλαδή, να είναι κανείς ε, δικαστής και διδητής σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο εύκολο. επιτρέπει ανεξάρτητο έλεγχο των διεκδικήσεων των καλλιεργητών και αυτοί μπορούν να επιλέξουν τον αυτόν που θα κρίνει. Ποιον ξεγελάμε. Δηλαδή δίνουμε το έδαφος Ευρώπης στη Μαλαισία. Ας το πούμε έτσι, καθαρά. Να μην χρονοτριβούμε, μην χάνουμε το χρόνο μας. Θεωρώ ότι αυτή η πρόταση θα σκοτώσει τα, τη γεωργία και τα βιοκαύσιμα που παράγονται στην Ευρώπη ε, και τα οποία θα μπορούσαν να είναι βιώσιμα αυτά, αυτά που είναι βιώσιμα και δεν οδηγούν στην ε, αποψήλωση των δασών. Να το πω ομά, ότι για αυτούς τους ε, δρόμους εγώ, για αυτούς τους λόγους εγώ θα προτείνω απόρριψη αυτής της κατεξουσιοδότηση πράξεως, ένσταση. Πριν δώσω το λόγο ξανά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας και να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτά που εφήγησαν. Ανεφερθήκατε σε αποδόσεις. Ξέρουμε ότι η απόδοση του φινικελαίου είναι πολύ υψηλότερη από ότι η απόδοση της σόγιας. Και το θέμα του κατοφλίου δεν είναι τόσο σαφές όπως το παρουσιάσατε. Με ένα όριο 10 όπως είπε ο Μπάς είναι χαμηλότερο από το όριο της σόγιας. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Σε αποφάσει που λάβαμε πρόσφατα για τα αυτοκίνητα, τα φορτηγάκια, τα βαρέα οχήματα. Χρειαζόμαστε μια ρύθμιση για τις χαμηλές ε, ε για να χαμηλώσουμε τις εκπομπές των οχημάτων και δεν το πετύχουμε μόνο με τα ηλεκτρικά οχήματα. Θέλουμε να, να γεφυρώσουμε τη διαφορά που υπάρχει και χρειάζεται ένα στοιχείο κατάλληλο και εδώ έχουμε σαν τέτοιο στοιχείο τα βιοκάψιμα. Έχετε προσμετρήσει τι ποσότητες προωθημένων βιοκαυσίμων χρειαζόμαστε για να πετύχουμε το στόχο. Να λάβουμε υπόψη τις αποφάσεις μας για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. θα είναι στα χέρια, είναι πολύ εύκολο αυτές οι μικρές εκμεταλλεύσεις να είναι υπό τον έλεγχο των μεγάλων εταιριών. Περιμένω τις απαντήσεις του κυρίου Φενστέιν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Είναι ένα θέμα το οποίο προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον. Ας ξεκινήσω με αυτό που είπατε στο τέλος, Πρόεδρε. Πράγματι, χρειάζονται κάποια βιοκαύσιμα στις μεταφορές και όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά πολύ περισσότερο στις αερομεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές, τις πλωτές μεταφορές και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε πολιτική για τα βιοκαύσιμα. Μια πολιτική που σαφέστατα καθορίζει το πώς σταδιακά μπορούμε να κινηθούμε προς βιοκαύσιμα δεύτερης και τρίτης ε, γενιάς και να αποφύγουμε τη χρήση βιοκαυσίμων που στην πραγματικότητα δεν μας κάνουν να πλησιάσουμε στους θεθέντες στόχους για την μείωση της χρήσεως και των εκπομπών άνθρακος. Αυτό είναι το ιστορικό, αυτό είναι το υπόβαθρο. Υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης ε, του θέματος του ILOG. Αυτό μας ζητήθηκε να κάνουμε. Σαφής εντολή που ε, δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθήσαμε να συμμορφωθούμε στο βαθμό των δυνατοτήτων μας. Και υπάρχουν κάποιες επιλογές που πρέπει να γίνουν. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε αφορά το φινικέλαιο. Είναι σαφέστατο ότι αν δούμε τα στοιχεία του φινικελαίου ηγείται, είναι κάτι ξεχωριστό όσον αφορά την επέκταση στη, στα αποθέματα και στην καλλιεργία το φινικέλαιο ε, έχει πρώτη θέση σε σχέση με άλλες ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται για τα βιοκάψιμα. Και για αυτό το λόγο μιλάμε για κάποιο μέτρο που θα αντιμετωπίσει το φινικέλαιο και θα μειώσει την ποσότητα του φινικελαίου που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοκαυσίμων ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο και σχετίζεται και με τα άλλα ερωτήματα που έθεσαν πολλοί ευρωβουλευτές που αφορούσαν τη σόγια. Όσον αφορά τη σόγια, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Τα ποσοστά αύξησης και επέκτασης της σόγιας είναι τέσσερις φορές χαμηλότερα από ό,τι είναι για το φινικέλαιο. Πολύ δύσκολο λοιπόν να κάνουμε τη σύγκριση και να πούμε ότι πρέπει στο ίδιο πλαίσιο να θέσουμε το φινικέλαιο και τη σόγια. Στο ερώτημα του κύριου Άικχαουτ, δηλαδή μήπως βάζουμε το όριο με τέτοιο τρόπο που με βολικό τρόπο δεν καλύπτουμε τη σόγια. Λέω όχι. Δεν κάνουμε κάτι τέτοιο που δεν είναι. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα βιοκαύσιμα που προωθούνται μέσω της οδηγίας είναι τα βιοκαύσιμα που οδηγούν σε πραγματικές οικονομίες. Και αν έχουμε μεγάλη επέκταση σε ε, εδάφη που παράγουν ζωοτροφές, δεν πετυχαίνουμε σωστά το στόχο μας. Και γι' αυτό βάλαμε το 10%. Θα μπορούσαμε να βάλουμε άλλα ποσοστά αλλά θεωρούμε ότι το 10% είναι το σωστό επίπεδο. Είναι πιο συντηρητικό από το 14% που αναφέρεται νομίζω στην οδηγία. Η έκταση ή μάλλον είναι η περιοχή κατά πόσο έχει οικονομία όσον αφορά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου ή όχι. Βάλαμε λοιπόν αυτό το όριο γιατί είχαμε το λόγο μας, τεκμηριωμένο. Ο κύριος Άικχαουτ ρώτησε τι αλλαγές μπορούμε να προτείνουμε ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα σχόλια που ακούσαμε. Και τα σημερινά και τα χθεσινά. Πολύ πρόημο να πούμε κάτι. Τώρα είναι η περίοδος των ανοιχτών διαβουλεύσεων. Μετά, όταν ολοκληρωθούν, θα δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Από όταν ετέθησε ισχύ οδηγία, παραμονές Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου, εργαστήκαμε άοκνα για να τηρήσουμε τις προθεσμίες που αναφέρατε κι εσείς. Δεν τα καταφέραμε απόλυτα, είμαστε ακόμα εδώ όμως. Εργαζόμαστε όσο πιο σκληρά γίνεται, διότι θα θέλαμε όλα αυτά να επιληθούν εντός της θητείας αυτού του Κοινοβουλίου και γι' αυτό και το Κοινοβούλιο στο κάτω-κάτω έθεσε αυτή την σύντομη αυτή προθεσμία. Ήταν εξαιρετικά σύντομο το χρονοδιάγραμμα για οποιαδήποτε κατοξισοδότηση πράξη σε οδήποτε τομέα νομοθεσίας και έχει ξεκινήσει η διαβούλευση. Συνεχίζεται και θα δούμε μετά τι αλλαγές θα προτείνουμε, αν υπάρχουν ευρείες επικρίσεις παρόμοιες με αυτές που ακούσαμε σήμερα και χτες. Για πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, στις λεπτομέρειες τώρα. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Υπάρχει μεγάλο κενό όπως κάποιοι διατείνονται. Δεν νομίζουμε. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις καθορίζονται σαφώς, πρέπει να είναι ανεξάρτητες μικρές εκμεταλλεύσεις. Αν όπως είπατε, στην πραγματικότητα είναι στη βιτρίνα ε, εικονικά είναι μικρές εκμεταλλεύσεις, ουσιαστικά δουλεύουν για κάποια μεγάλη επιχείρηση. Μιλάτε για μίσθωση. Μιλάτε για μίστοση. Εάν κάποιο είναι μικρό εκμεταλλευτή, μικρό καλλιεργητή και μισθώνει η γη, αυτό πώ λειτουργεί. Η μίσθωση, η περίπτωση τη μίσθωση και όχι διοκτησία. Με τα χαρά να μπούμε σε μια συζήτηση. Μου λέγουν ότι στο νομικό κείμενο έχουμε ρήτρα διαφύλαξη. Σύμφωνα με την οποία αν είσαι μικρό καλλιεργητή, αλλά μόνο κατόνομα και όχι στην πραγματικότητα, τότε δεν μπορείς να ε, τύχη αυτή τη εξαίρεση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, για τους μικρούς καλλιεργητές. Το μόνο που δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι η οικονομική συμπληρωματικότητα όσον αφορά τα κριτήρια. Όλα Τα κριτήρια πρέπει να πληρούνται. Πρέπει να αποδείξουν συμμόρφωση με τα κριτήρια ε, βιωσιμότητας. Δεν είναι δίκιο να λέει κανείς ότι εδώ είναι η συνηθισμένη προσέγγιση. Όχι. Δεν αποτελεί αυτή η προσέγγιση συνέχεια της χρήσης του φινικελαίου για παραγωγή βιοκαυσίμων ή χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σταδιακή εξάλληψη που προβλέπεται, καθορίζεται σαφώς μέχρι την περίοδο του 2030. Αυτό τα αποφάσισαν ξεκάθαρα οι συνομοθέτες έλεγχος. Βάσει αυτών των κριτηρίων είναι ίδιος έλεγχος όπως και για τα κριτήρια βιωσιμότητας. Αναφέρονται στη σημερινή οδηγία, στην ισχύουσα οδηγία. Νομίζω ότι λειτουργούν καλά, είναι αξιόπιστα τα κριτήρια, τα όλα πλαίσια που έχουμε, τα σχήματα που έχουμε, τα συστήματα για αναγνώριση, για συμμόρφωση με τα κριτήρια. Είναι καλά, είναι καλοί μηχανισμοί. Δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης. Να θεωρήσουμε ότι διαπράττονται απάτες. Μιλάμε για ανεξάρτητο έλεγχο. Βέβαια τα κριτήρια που ανα γιατί αναφέρθηκαν και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κριτήρια δεν επεκτείνονται στο κατά πόσο υπάρχουν παραβιάσεις ή προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την παραγωγή των ζωοτροφών. Μπορεί να υποβάλλονται καταγγελίες και αναφορές πέραν των κριτηρίων, αλλά δεν αποτελεί αυτό ο τομέας ε, κριτήριο. Ελπίζω να απάντησα στι περισσότερε ερωτήσεις. Τώρα, όπως ε, προανέφερα, είμαστε στη δημόσια διαβούλευση Είμαστε σε επαφή με πολλούς ε, εμπλεκομένους φορείς, παραγωγούς και καταναλωτές. Άκουσα προτάσεις που είπαν ότι μάλλον κάποιοι διατείνονται ότι έχουμε πλησιάσει κάποιες χώρες παραγωγούς. Ακούσαμε κάποιες, αλλά ακούμε όλους τους πάντες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε πολύ ανοιχτοί. Διεξάγονται ειλικρινείς ε, συζητήσεις και με ΜΚΟ και με τις παραγωγές χώρες αυτός είναι σωστός τρόπος διεξαγωγής αυτών των συναλλαγών. Γνωρίζουμε όλες τις επικρατούσες απόψεις για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ εκ νέου που με ακούσατε. Εάν έχω ξεχάσει κάποια ερώτησή σας, με τα χαράς να σας απαντήσω σε μια διαδικασία που θα ακολουθήσει αυτό το στάδιο των ρωταπαντήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε και ευχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλή τύχη στις προσπάθειές σας για βελτίωση του θέματος αυτού. Ενημέρωση λοιπόν για την επόμενη συνεδρίαση 26-27 Φεβρουαρίου. 27 Φεβρουαρίου από 9 το πρωί θα ξεκινήσουμε από 9 μέχρι 12.30 λοιπόν και από 2.30 μέχρι 6.30 το απόγευμα. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.